Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έντιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το θέμα το οποίο γύρεται από αυτή την ερώτηση αφορά πράγματι τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία είναι κεντρικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι και ο κύριος γνώμονας εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα σα διαβεβαιώσω ότι είναι απόλυτα προσφυλωμένη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα ανθρώπινα δικαιώματα και στις κέρυε συμβάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας μέσα στους οποίους αναφέρεται και το θέμα της απαγόρευσης της ε, καταναγκαστικής εργασίας. Γνωρίζετε συγχρόνω πόσο λεπτό είναι το θέμα αυτό και γνωρίζετε πόσο λεπτή είναι και η σχέση μα με την Ταϊβάν. Γνωρίζουμε ότι το σύστημα των Λαογκάι είναι τμήμα της προσπάθειας της Κίνας να γίνει μια σύγχρονη και ανεπτυγμένη κοινωνία. Η διατήρηση αυτού του συστήματος είναι απόλυτα συμβατή με τις δεσμές που έχει αναλάβει η Κίνα στον τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων και την δήλωσή της ότι θα ακυρώσει την Διεθνή Σύμβαση για τα πολιτικά και αστικά δικαιώματα που υπέγραψε πριν από 12 χρόνια, μονογράφησε πριν από 12 χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει πράγματι ένα πρόβλημα, διότι τα αγαθά που παράγονται στα ΛΑΟΓΚΑΙ κάτω από αυτέ τις καταδικαστέ συνθήκε μπορεί να εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι πολύ δύσκολο να μπορέσουμε με επακριβή τρόπο να καθορίσουμε ποια αγαθά που εισάγονται από την Κίνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν παραχθεί σε ΛΑΟΓΚΑΙ απαντών σε προηγούμενες ερωτήσεις από τη πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της κοινωνίας των πολιτών και των φορέων της κοινωνίας των πολιτών, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει αυτό το θέμα με συνέπεια και κατ' επανάληψη με την, στις συζητήσεις μας με την Κίνα τα τελευταία χρόνια, ιδίως μέσα στα πλαίσια του ε, εξαμηνιαίου διαλόγου ανθρωπίνων δικαιωμάτων με την Κίνα. Στα πλαίσια αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υπογραμμίσει ότι το σύστημα Λαογκάι παραβιάζει πολλά άρθρα της Διεθνούς Σύμβασης για τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα και ιδίως το άρθρο 8 το οποίο απαγορεύει την υποχρεωτική ή καταναγκαστική εργασία καθώς και το άρθρο 9 το οποίο λέει ότι κανείς δεν θα πρέπει να φυλακίζεται χωρίς προηγούμενη δίκη. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοίμησε να χρησιμοποιήσει μια θετικής, μια, μια προσέγγιση θετικού διαλόγου με την Κίνα αντί να καταφύγει σε μια απαγόρευση εισαγωγών. Αλλά θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν και όρια σε αυτή την προσέγγιση που μέχρι τώρα δεν οδήγησε σε κάποια ουσιαστική αλλαγή στην πολιτική της Κίνας σε ό,τι αφορά τα Λάο Γκάι. Πρέπει να αναγνωρίσουμε επίσης ότι η Κίνα δεν είναι η μόνη χώρα όπου τίθεται το θέμα της εργασίας των κρατουμένων σε φυλακές. Η Κομισιόν επομένως έχει ανοιχτό πνεύμα στο να ε, αναθεωρήσει την άποψή της για το ερώτημα αυτό, να, το αναθεωρήσει τα στοιχεία και να ασκήσει πίεση σε όλες τις χώρες οι οποίες χρησιμοποιούν εργασία κατουμένων σε φυλακές, παραβιάζοντας έτσι θεμελιώδεις αρχές ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συμβάσεις της διεθνούς κοινότητας και του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας. Αυτό θα πρέπει να γίνει με ένα οριζόντιο τρόπο και δεν θα πρέπει να περιορίζεται μονάχα στην Κίνα. Χαιρετίζουμε λοιπόν τις απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο για τα θέματα αυτά και θα σας κρατήσουμε ενήμερους για τις περαιτέρω εξελίξεις. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε. Κύριε Πίτροπε, ακολουθούν οι ομιλητές εξορμώσεις των πολιτικών ομάδων. Ο κύριος Γκάλερ για 1,5 λεπτό έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλό είναι να κάνουμε αυτή τη συζήτηση στην ίδια Ολομέλεια όπου συζητήσαμε και για την διάσκεψη κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας. Υπάρχει και μια εμπορική αλλά υπάρχει και μια πτυχή ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα θέματα αυτά. Στη δεύτερη εγώ θα επικεντρωθώ η εργασία η καταναστατική στα ΛΑΟΚΑΟ έχει σύνθημα εργασία η οποία οδηγεί στην πρόοδο. Όλα αυτά γίνονται σε συνθήκε οι οποίε είναι απόλυτα απαράδεκτε και όχι και αποδεκτέ για του εταίρου τη Ευρωπαϊκή τη Κίνα. Αντιβαίνουν στα ανθρώπινα δικαιώματα και όλε τι ε, υποχρεώσεις που έχει συνάψει η Κίνα με το να υπογράψει τη Σύμβαση για τα, ανθρώπινα, για τα πολιτικά και αστικά δικαιώματα. Είναι κάτι λοιπόν το οποίο το έχουμε καταδικάσει όλοι. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι φυλακές Λαουγκάι εμφανίζονται ως εμπορικές εταιρείες και με τον τρόπο αυτό αποκρύπτουν τον πραγματικό τρόπο λειτουργίας τους. Στις Ηνωμένε Πολιτείε έχει υπάρξει μία απαγόρευση της εισαγωγής προϊόντων από τέτοιες, ε, ε, από τέτοιες πηγές και έχουν εφαρμόσει αυτή την απαγόρευση κατά αυτών των επιχειρήσεων. Λέτε ότι είναι πολύ δύσκολο να ξέρουμε από πού προέρχονται αυτά τα προϊόντα, αλλά τα ονόματα αυτών των επιχειρήσεων που είναι πράγματι λαογκάι και είναι στατόπεδα κρατουμένων, είναι γνωστά αυτά τα προιοντα αλλα τα ονοματα αυτων των επιχειρησεων που ειναι πραγματι λαογκαι και ειναι τοπεδα κρατουμενων ειναι γνωστα αυτα τα ονοματα Οι ΗΠΑ έχουν ήδη συγκεκριμένη εμπειρία για τι εταιρείε αυτέ που παράγουν τέτοια προϊόντα. Επομένω το ερώτημα είναι αν είσαστε έτοιμοι να λάβετε υπόψη τον κατάλογο αυτών των επιχειρήσεων και να προβείτε σε ανταλλαγή εμπειριών με τι Ηνωμένε Πολιτείε, ώστε με τον τρόπο αυτό να μπορέσει να γίνει κάτι για να αντιμετωπιστούν αυτά τα προϊόντα. Και η τελευταία ερώτηση μου είναι το εξή. Αν θα ζητήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση από την Κίνα ο ειδικό αντιπρόσωπο των Ηνωμένων Εθνών για την ε, για τα βασανιστήρια να επισκεφτεί περιοχές όπως το Χσισιάν και το Θιβέτ. Ευχαριστώ. Η κυρία Κάλεμπαχ για τρία λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών ενδιαφέρεται ιδιαίτερα ε, να συνεχιστούν οι επικοδομητικές σχέσεις με την λαϊκή δημοκρατία της Κίνας. Όμως, η απάντησή σας με απεγοήτευσε. Δηλαδή, δεν είπατε απολύτως τίποτα το ξεκάθαρο. κρυφτήκατε λίγο πίσω από το γεγονός ότι είναι δίθεν δύσκολο να θέσει κανείς τα τέτοια θέματα. Αλλά αυτό <clears throat> δεν είναι δικαιολογία. Οι Ηνωμένε Πολιτείε, για παράδειγμα, βρήκαν ξεκάθαρε λύσει για το ίδιο θέμα. Ο θετικό ισολογισμό των εμπορικών σχέσεων με την Κίνα, μακάρι να υπάρχει τέτοιο, δεν μπορεί ωστόσο να είναι λόγο για να <clears throat> κλείνουμε τα μάτια απέναντι σε βαριέ παραβιάσει των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Άλλωστε θα ωφελήσει και την ίδια την Κίνα και του εκπροσώπου της οι οποίοι, και τους εκπροσώπους της όπως λέω, οι οποίοι σίγουρα προσπαθούν να φέρουν μια ισορροπία ανάμεσα <clears throat> στις ε, παράκτιες περιοχές οι οποίες ε, βλέπουν να αυξάνεται διαρκώς το εισόδημά τους και τις εσωτερικές βασισμένες στην αγροτική οικονομία περιοχές οι οποίες ε, τα πηγαίνουν πολύ χειρότερα. Δεν λέω ότι πρέπει να απογορευτεί η εισαγωγή των προϊόντων αυτών. Υπάρχουν όμως πολλά μέτρα που μπορούν να ληφθούν. Υπάρχει η δυνατότητα να υποδείξουμε στις ευρωπαϊκές μας επιχειρήσεις ποια προϊόντα φέρουν τις ε, επωνυμίες των επιχειρήσεων αυτών που είναι στην πραγματικότητα συγκάλυψη του γεγονότος ότι τα προϊόντα θα παράγονται στα Λαογκάι πρέπει να εμείνουμε ε, ε, και να επιμείνουμε ώστε τα, δικαιώματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα να διατηρούνται, να τηρούνται μάλλον, να γίνονται σεβαστά. Εγώ είμαι και εκπρόσωπο ε, των καταναλωτών και καταναλωτών που θέλουν να έχουν την βεβαιότητα όταν αγοράζουν κινέζικα προϊόντα ότι δεν πρόκειται για προϊόντα καταναγκαστική εργασία. Ήδη η ευαισθητοποίηση προϊόντων που προέρχονται από παιδική εργασία είναι σημαντική και έχουμε λάβει μέτρα. Αναμένω λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκεκριμένε προτάσει σχετικά για παράδειγμα με μια σφραγίδα ποιότητας ε, των προϊόντων και διάφορα άλλα τέτοια μέτρα και ελπίζω και εύχομαι να συνεχιστεί ο επικοδομητικός διάλογος με την Κίνα. Βλέπω και από πλευράς της κινέζικης κυβέρνησης να υπάρχει η θέληση να συνεχιστεί ο διάλογος. Και η Κίνα ενδιαφέρεται να βελτιώσει την κατάσταση των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην χώρα αυτή. Και διότι οι εμπορικές σχέσεις είναι τόσο σημαντικές. Ευχαριστώ. Ο κ. Γκέρενς. Πρόεδρε, πάνω από χίλια στρατόπεδα σύμφωνα με εκτιμήσεις ε, ΜΚΟ Τρία με πέντε εκατομμύρια άνθρωποι είναι φυλακισμένοι με την υποτιθέμενη κατηγορία ε, στην ασφάλεια του κράτους. Ε, ωστό, ακόμα και αν δεν είναι εξαντλητικός ο κατάλογος αυτός, είναι πολύ ανησυχητικός. Η αντίδραση της διεθνούς κοινότητας, ωστόσο, παραμένει πολύ δειλή. Αυτό που περιμένουμε από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να μας πει με τριπαθή βήματα, ωστόσο που θα είναι πιθανόν να οδηγήσουν όλους τους εμπορικούς εταίρους της Κίνας να κρατήσουν σταθερή στάση ώστε να επιτύχουν σημαντικές υποχωρήσεις. Έχουμε ήδη δημιουργήσει task force για λιγότερο σημαντικά θέματα. Ευχαριστώ κύριε Ένα λεπτό, Μιγκάλσκι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, και εγώ συμπαρατάσσομαι με εκείνους που λέγουν ότι η ομιλία σας μας απογοήτευσε. Το θέμα αυτό θα πρέπει να είναι θέμα κλειδί για μας. Στα στρατόπεδα Λαογκάη ζουν 7 εκατομμύρια άνθρωποι που διώκονται λόγω θρησκευτικών ή πολιτικών πεπιθήσεων. Είμαστε λοιπόν ηθικά και πολιτικά υποχρεωμένοι να αντιταχθούμε. Εμείς έχουμε την εντύπωση ότι αυτό το σύστημα στρατοπέδων ε, θυμίζει τα σοβιετικά γκουλάγκ. Και το όνομα το ίδιο. γκάι σημαίνει αλλαγή μέσω της εργασίας. Πράγματα δηλαδή που έγραφαν και τα γερμανικά στρατόπεδα συγκεντρώσεως της ναζιστικής εποχής, όπως τα Auschwitz, επάνω από την είσοδό τους. Αυτά τα πράγματα Αυτά τα θέματα θα πρέπει να είναι θέματα κλειδί στι συζητήσει μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας. Σας προτρέπω κύριε Επίτροπε να θέσετε το θέμα διαρκώς, να το θέτετε διαρκώς σε κάθε συζήτηση με, με Κινέζου Κύριε Η κυρία Βεργιά, λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όλοι γνωρίζουμε τι γίνεται με την δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κίνα. Μιλήσαμε για την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονία και στι δύο περιπτώσει με ένα κοινό σημείο. Ότι δηλαδή ο οικονομικό ρεαλισμό επικρατεί. Γιατί η Κίνα καταρχήν για όλου όσου δικούν την Ευρώπη είναι μια μεγάλη αγορά. Ε, θα μπορούσαν να μας κλείσουν τις, ε, τα σύνορα. Και δεν έχει σημασία που η πολιτική καταπίεση και καταστολή είναι η ίδια. Εγώ δεν ξέχασα τα θύματα της Tiananmen. Δεν ε, ξεχνώ όλους αυτούς που σαπίζουν στη φυλακή ή σε στρατόπεδα εργασίας και που με τη ζωή τους ε, πληρώνουν τον αγώνα για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τα λαογκά είναι ένα φρικτό μήνυμα, δείγμα του τι συμβαίνει στην Κίνα. Κύριε Πίτροπε, μην κρύβεστε πίσω από τεχνικές δικαιολογίες και μην προσπαθείτε πια να συνοηθείτε με την κινέζικη κυβέρνηση. Ξέρετε ε, πώς ε, λαμβάνουν υπόψη τους αυτές τις συζητήσεις. Είναι υποχρεωτικές ε, συναντήσεις για αυτούς απλώς. Δεν έχουν πει τίποτα συγκεκριμένα. και μην κρύβεστε πίσω από το γεγονός ότι υπάρχουν και αλλού στρατόπεδα εργασία. Η Κίνα εξυγχρονίζεται μας λέτε. Εγώ θα έλεγα ότι όχι, δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δεν είμαι υπέρ τον είπα, όχι. Αλλά αυτό που κάνουν είπα είναι αυτό που θα έπρεπε να κάνουμε. Ξέρουμε να συνεργαστούμε μαζί τους, ε, ακόμα και με την περιφρόνηση των Ευρωπαίων πολιτών. Γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε και όταν θέλουμε να τηρηθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κύριε Επίτροπε, Πότε η Ευρωπαϊκή Ένωση θα απαγορέψει την εξαγωγή προϊόντων από τα στρατόπεδα Λαογκάη. Ευχαριστώ κυρία Βερζία για ένα λεπτό τώρα ο συνάδελφος Σοντάνα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Τα όσα μας είπατε δεν, είναι, δεν ήταν αυτά τα οποία προσδοκούσαμε. Περιμέναμε να είσαστε πιο αποφασιστικός. Δεν μπορούμε να δεχόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα να ε, υποκύπτουν στην οικονομία. Υπάρχουν εκατομμύρια στα λαόγκα, εκατομμύρια άτομα των οποίων τα δικαιώματα καταπατώνται και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτό είναι πρόβλημα και για την ευρωπαϊκή οικονομία, διότι τα προϊόντα που φτάνουν στις αγορές μας δημιουργούν αυτόν τον αθέμητο ανταγωνισμό και προκαλούν μεγαλύτερη κρίση στην Ευρώπη. Είναι ζήτημα ανταγωνιστικότητα, ντάμπινγκ κλπ. Όλα αυτά λοιπόν μα κάνουν να καταλάβουμε πω μολονότι η κυβέρνηση του Πεκίνου έκανε και είπε κάποια πράγματα, δυστυχώ το αποτέλεσμα δεν το βλέπουμε. Τα λογά συνεχίζουν να υπάρχουν και δυστυχώ εκατομμύρια άνθρωποι που αποτελούν και μειονότητε στη χώρα αυτή βλέπουν τα δικαιώματά τους να καταπατώνται. Εύχομαι πως η λογική της διπλωματίας και της ε, διαβούλευσης θα υπερισχύσουν και η Ευρώπη θα μπορέσει να απαγορεύσει την εισαγωγή αυτών των προϊόντων λαογκάι ακόμα και στις ΗΠΑ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ακούσουμε τώρα τους υπόλοιπους ομιλητές. Για 1,5 λεπτό ο κύριος Κάσπαρη. Κύριε Πρόεδρε, Κυρίε και κύριοι, όλοι γνωρίζουμε πως πίσω από τα λαόγκα κρύβεται ένα απαράδεκτο σύστημα στρατοπέδων εργασία στην Κίνα και μόνο η ύπαρξή του είναι απαράδεκτη. Αλλά όταν χρειάζεται να φανταστώ πω κάποια προϊόντα παράγονται εκεί πέρα, είναι και στα μαγαζιά μα, πλέον η κατάσταση είναι αφόρητη. Δεν φτάνει δηλαδή που αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται στο στρατόπεδο εργασία, αλλά να κερδοσκοπεί βάρο του και η κινέζικη κυβέρνηση είναι απαράδεκτο οπωσδήποτε εμένα θα μου κόβονταν οποιαδήποτε όρεξη αν γνώριζα πως ε, έχω μπροστά μου προϊόντα που παρήχθησαν ε, εκεί πέρα. Οπότε πρέπει επιτέλους κύριε Επίτροπε να δει η Κομισιόν πρώτα απ' όλα σε ποιες άλλες χώρες ε, παράγονται αυτά τα προϊόντα σε φυλακές και έρχονται σε εμάς. Δηλαδή ασχοληθείτε μία φορά με ένα πρόβλημα σωστά, λύστε το και μετά περάσει το επόμενο. Ζητώ από Κομισιόν και Συμβούλιο επιτέλους να διασφαλίσουν πως τα προϊόντα από αυτά τα στρατόπεδα πλέον δεν θα μπορούν να αγοραστούν. Δεν θέμε αυτά τα προϊόντα στην Ευρώπη. Οι ΙΠΑ βρήκαν έναν τρόπο να τα απαγορεύσουν Ζητώ λοιπόν από την Κομισιόν αυτά τα προϊόντα τα βαμμένα με αίμα να μην ξανάρθουν σε εμάς. Εύχομαι και επιθυμώ καλή συνεργασία με την Κίνα, αλλά πλέον αυτά τα προϊόντα πάντα θα μοδρώνουν αυτή τη συνεργασία. Ευχαριστώ κύριε Κασπάρη. Η κυρία Μάισνερ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, είπατε πως τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι θεμελιώδης αξία της Ένωσης. Τον προηγούμενο Δεκέμβριο εγκρίναμε όλο περηφάνεια τη συνθήκη της Λισαβόνας, στην οποία βεβαίως υπάρχει και η χάρτα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και είναι σωστό αυτό το οποίο είπατε, πως θα πρέπει να υπρασπίζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα παντού και να προσανατολιστεί ανάλογα και η οικονομική μας δραστηριότητα. Ήδη όμως υπόθηκε πως ε, με τα προϊόντα από το Λαογκάι δεν ξέρετε ποιο παράγεται πού. Εγώ έχω ένα, προϊόν, ένα βιβλίο εδώ πέρα που αναφέρει ποιο προϊόν προέρχεται από ποιο στρατόπεδο κτλ. Υπάρχει το Ίδρυμα Ερευνών για τα Λαουγκάι και νομίζω και ο κύριος Πέτρι Μίλλερ νομίζω μπορεί να απευθυνθεί στον κύριο Ντεχούχτ για να του ζητήσει να δει τι γίνεται με τον ειδικό απεσταλμένο του ΟΗΕ για τα στρατόπεδα αυτά εργασία. Και δηλαδή έχουμε φτάσει στο σημείο η ΙΠΑ να είναι πιο θαραλέες από εμά και να έχουν απαγορεύσει αυτά τα προϊόντα. Πρέπει τέλος να κάνει κομισιόν αυτό το οποίο μα προσχέθηκε. Ευχαριστώ κύριε Μάισνερ. Ο κύριος Προβέρα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε να αναφέρω μερικά στοιχεία πάνω από χίλιαντα στρατόπεδα λαϊκά, τα οποία είναι ε, εξακριβωμένα και πάνω από 5.000 5 εκατομμύρια κρατούμενοι από το 59 και ε, Λαογκάι ένα σύστημα φυλάκισης από το πλέον καταπιεστικά στον κόσμο βασισμένα στο μοντέλο των γκουλάκ της Σοβιτικής Ένωσης για να τιμωρήσουν τους ε, αντικαταστατικούς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, με πολλά, έχει πολλά προβλήματα να αντιμετωπίσει τα εισαγόμενα προϊόντα από την Κίνα διότι δεν, υπάρχει καμία προστασία των εργαζομένων. Τώρα θα δεχθούμε επίσης και προϊόντα τα οποία κατασκευάζουν πολιτικοί κρατούμενοι είμαστε, είναι σαν να συμβάλλουμε κι εμείς σε αυτό το έγκλημα. Διαφορετικά κύριε Επίτροπε θα δώσουμε την εντύπωση ότι ασκούμε κριτική προς τις μικρές χώρες αλλά είμαστε πολύ επιφυλακτικοί και προσεκτικοί απέναντι σε μεγάλες χώρες όπως η Κίνα. Η επόμενη διάσκεψη του Οκτωβρίου θα είναι μια ευκαιρία να θίξουμε το πρόβλημα αυτό. Εύχομαι κύριε Επίτροπη η ευκαιρία αυτή να μην πάει χαμένη και να έρθετε να μας πείτε νέα καλύτερα. Ευχαριστούμε κύριε Προβέρα. Συνάδελφος ο κύριος Πρέντα για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το άρθρο 11 της Οικουμενικής Διακήρυξης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προβλέπει το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη. Είναι προφανές ότι στα στρατόπεδα Λαογκάη παραβιάζεται αυτό το δικαίωμα. Όπως είπαν πολλοί συνάδελφοι, όχι μόνο δεν δικάζουν δίκαια, αλλά υποβάλλουν σε βασανισμό τους κρατούμενους, σε καταναγκαστική εργασία, σε ξεφτελιστική μεταχείριση ουσιαστικά σε δουλεία γιατί τους υποχρεώνουν να εργάζονται ακόμη και 24 ώρες 24 ώρα μερικές φορές, εργοστάσια, ορυχεία κτλ. Επίσης υπάρχουν, υπάρχει κακομεταχείριση, ξυλοδαρμοί, βιασμοί σε αυτά τα στρατόπεδα Λαο Γκάι και οι κρατούμενοι δεν δικαιούνται καν υγειονομική περίθαλψη ή φάρμακα. Η εισαγωγή τέτοιων προϊόντων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να απαγορευτεί ολοσχερός. Εγώ αυτό πιστεύω και ελπίζω να παρακολουθήσει την σωστή τήρηση αυτής της απαγόρευσης Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως ζήτησαν και άλλοι συνάδελφοι. Και εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε κάθε ευκαιρία στις ε, διασκέψεις υψηλού επίπεδου με τους ε, Κινέζους ομολόγους μας και να ζητήσουμε να απαγορευτεί αυτό το σύστημα των στρατοπέδων. Κυρία Μοσκαρδίνη, για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όποιος ε, ακολουθεί τον ε, νόμο του Μαμονά δεν ε, θα, δεν θα πρέπει να ακολουθούμε αυτόν τον νόμο διότι με αυτόν τον τρόπο συμβάλλουμε στο να συνεχίζουν να καταπιέζονται άτομα και να εισάγουμε στην Ευρώπη ματωμένα προϊόντα. Δεν νομίζω λοιπόν ότι το ηθικό μας ε, ζήτημα θα μπορέσει να μας βοηθήσει να επιλύσουμε τα προβλήματα αυτά, διότι δεν έχουμε ακόμα μέτρα, μέτρα για να απαγορεύσουμε αυτές τις αγωγές και συνεχίζουμε διαπραγματεύσεις με τη λαϊκή δημοκρατία της Κίνας, μόνο ότι γνωρίζουμε πολύ καλά το τι πράττει η Κίνα και το ποια είναι η προέλευση αυτών των προϊόντων φοβούμε ότι το ηθικό θέμα δεν ε, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ευρώπη. Γι' αυτό λοιπόν το Κοινοβούλιο μας ε, κάνει μια έκκληση προκειμένου να επανέλθετε στο θέμα με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και να αντιμετωπίσετε με την Κίνα με τρόπο ξεκάθαρο και σαφή το πρόβλημα αυτό. Εν τω μεταξύ η Ευρώπη επειδή φοβάται και την οικονομική της κατάσταση, τουλάχιστον θα πρέπει να κινηθούμε για να έχουμε το συντομότερο έναν κανονισμό για τον ονομασία προέλευσης και έτσι μπορούμε να πούμε ότι στην κοινωνική κυβέρνηση ότι αν δεν απαγορευτεί η κατασκευή αυτών των προϊόντων από κρατούμενος και η εξαγωγή αυτών όλα τα προϊόντα που θα πρόκειται από την Κίνα για μας ε, θα θεωρηθεί ως προϊόν το οποίο φέρει ε, μαζί του και το αίμα. Ευχαριστώ. Στο τελευταίος από τους ε, ομιλητές, ο κύριος Κέλλαμ για μισή λεπτό. Κύριε Επίτροπε, δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι ένα σημαντικό τμήμα της οικονομικής ανάπτυξης Κίνας οφείλεται στην οικονομία των φυλακών. Και μάλιστα ε, τα στρατόπεδα και οι μαζικές κρατήσεις ισχύουν από το 49 και ήταν το σημαντικότερο ε, ε, μέσο καταπίεσης. 15 ε, εκατομμύρια ήταν συνολικά οι πολιτικοί κρατούμενοι και 5 εκατομμύρια από αυτούς βρίσκονται σε κρατικές φυλακές. Και μάλιστα η καταναγκαστική εργασία στα στρατόπεδα της Κίνας είναι ουσιαστικά ένα κοινό μυστικό. Και πολλά προϊόντα παράγονται στα στρατόπεδα αυτά. Και μάλιστα εν ώψη της διάσκεψης κορυφής που θα έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Κίνα, σας ερωτώ κύριε Επίτροπε, είστε έτοιμος να εφαρμόσετε την αρχή αμοιβαιότητας του Προέδρου Βαν Ρόμποϊ στη σχέση μας με την Κίνα. Θα πρέπει να ασκήσουμε πιέσεις προς την κατεύθυνση αυτή υπάρχει καμία συνεργασία με τις Αμερικανικές Αρχές σε ό,τι αφορά την ανείχνευση προϊόντων από στρατόπεδα Λαογκάη. Ρίξτε καμιά ματιά σε προηγούμενα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είναι υπέρ τη ολοσχερού ε, απαγόρευση προϊόντων από τα στρατόπεδα Λαογκάη στην Ευρώπη. Και επιμείναμε η πρόοδο των διαπραγματεύσεων με το Πεκίνο να εξαρτηθούν από την προηγούμενη επικύρωση από την Κίνα των χαρτών του ΟΗΕ και τη Διεθνού Οργάνωση Εργασία. Και τι θα γίνει σε περίπτωση που αρνηθούν κάτι τέτοιο οι Κινέζικε αρχέ. Νομίζω ότι σε όλε αυτέ τι ερωτήσει δικαιούμαστε μία απάντηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κέλλαμ, πρώτος ομιλητής στη διαδικασία και έτσι για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το να στέλνονται οι άνθρωποι σε στρατόπεδα εργασία γιατί σκέφτονται διαφορετικά από το καθεστώς είναι βεβαίως κάτι το οποίο προσβάλλει τον, τον ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Αναχρονισμοί που δεν έπρεπε να υπάρχουν στον 21ο αιώνα πουθενά στον κόσμο και απογοήτευμε Απογοητεύομαι γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν κατάφερε να κάνει τίποτα καλύτερο στην περίπτωση της Κίνας παρά το ότι ήξερε και δεν έχει κάποια βήματα για το πώς η περαιτέρω συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, Κίνας θα προχωρήσει. Όταν υπάρχουν site, όταν υπάρχουν βιβλία που αναφέρουν τα προϊόντα αυτά και από πού προέρχονται, γιατί δεν τα ξέρετε εσείς, κλείνετε τα μάτια εδώ πέρα. Ε, εσείς λοιπόν και οι Κομισιόν είστε συνυπεύθυνοι για τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι έχουν φυλακιστεί με αυτές τις δίκες θέατρο. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Το κράτος δικαίου είναι βασική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ντρέπομαι ως Ευρωβουλευτής για αυτά τα οποία ακούμε σήμερα, αλλά από την άλλη χαίρομαι για το ότι όλοι διακομματικά θέλουμε αυτή την αρχή του κράτους δικαίου και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κάσλε. Ο κύριος για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, οι συνάδελφοι είπαν πως είναι κάτεπίγον για τα ανθρώπινα δικαιώματα να σταματήσει η εισαγωγή αυτών των προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εγώ θεωρώ πως υπ' αυτές τις απάνθρωπες συνθήκες ε, παράγονται προϊόντα πρέπει να δούμε το εάν μπορούμε να κινήσουμε και μια διαδικασια διαδικασία anti-dumping με τις τιμές αυτές. Επίσης θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι ως Ευρωπαϊκή Ένωση, ανεξαρτήτως των εμπορικών θεμάτων. Δεν είναι αποδεκτές αυτές οι συνθήκες που επικρατούν σε αυτά τα στρατόπεδα. Δεν είναι το θέμα τα προϊόντα, είναι το πώς ζουν οι άνθρωποι, οι κρατούμενοι εκεί πέρα, οι οποίοι δεν έχουν καμία εγγύηση του κράτους δικαίου. Πρέπει να το πω, ξεκαθαρίσουμε αυτό στην ε, Κινέζικη Δημοκρατία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Λίχτενμπέργκερ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Επίτροπε, είπατε πως είναι ευαίσθητες οι σχέσεις με την Κίνα. Ναι, αλλά θεωρώ πως μεταξύ εταίρων οι οποίοι εμπορεύονται μεταξύ τους, ε, που συνεργάζονται σε παγκόσμιο επίπεδο, νομίζω είναι αναγκαίο ο καθένας να μην τονίζει μόνο τις αρχές του, αλλά να βγάζει και τα απαραίτητα αποτελέσματα στις διαπραγματεύσεις. Αλλιώς θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και για υποκρισία, δηλαδή όταν ο ένας ασκεί κριτική στην κατάσταση αυτά στα στρατόπεδα, που συμφωνώ βεβαίω, αλλά από την άλλη επιτρέπει να έρχονται τα προϊόντα αυτά στην αγορά του. Είναι θέμα ευρωπαϊκής αξιοπιστίας. Ότι δεν πρέπει δηλαδή μόνο να μιλάμε, αλλά να δράσουμε κιόλας. Γι' αυτό θεωρώ, επειδή σεβόμαστε βεβαίως την Κίνα, όταν και εμάς μας βλέπει τόσο υποκριτές δεν θα μας πάρει τόσο πολύ στα σοβαρά όταν ε, υποβαθμίζουμε τις αξίες μας έναντι του εμπορίου. Ευχαριστώ κύριο Τάνοκ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η Κίνα είναι ουσιαστικά ε, οικονομικός καταλήτης και θαύμα, αλλά είναι και μια αποτρόπαια κομμουνιστική χώρα. Μάλιστα, Βλέπουμε πως ε, χρησιμοποιείται και τα αναγκαστική εργασία στα στρατόπεδα που στέλνει αντιρρησίε συνείδηση πολιτικούς κρατουμένους, ε, οπαδούς της Φαλούν και υποτίθεται ότι στέλνονται εκεί για σοφρονισμό και για αναμόρφωση. Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες ε, ότι χρησιμοποιούνται οι κρατούμενοι για εξαγωγή οργάνων για δωρεά, βασανίζονται και πολλές φορές ε, υπάρχει και ένα άλλο θέμα που είχα θίξει στο παρελθόν και προς τον κύριο, στον Επίτροπο Μάντερσον, είναι αυτή η ανησυχία ότι τέτοιου είδους καταναγκαστικά στρατόπεδα ε, παράγουν αγαθά. Για παράδειγμα, λαστιχένιες μπότες που φτάνουν στις ευρωπαϊκές αγορές. Βέβαια, ε, είναι δύσκολο, ήταν δύσκολο μέχρι στιγμής για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εντοπίσει τέτοια προϊόντα και να αποδείξει την προέλευσή τους. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό, κύριος Πάσκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Τα Λαογκάι, τα στρατόπεδα αυτά εμφανίστηκαν μετά την Κομμουνιστική Επανάσταση του 1948 Έκτοτε έχουν περάσει από αυτά γύρω στα 50 εκατομμύρια Κινέζοι και μόνο μισή γύρισαν σπίτια τους. Σύμφωνα με το Ίδρυμα Έρευνας για τα Λαογκάι, αυτή τη στιγμή υπάρχουν γύρω στα 1.700 τέτοια στρατόπεδα και εκεί πέρα φτάνει κανείς και αποστέλλεται χωρίς ε, καν δικαστική απόφαση, παρά μόνο με απόφαση της αστυνομίας. Ναι, δεν βλέπουν αυτοί οι άνθρωποι τους συγγενείς τους ε, παρά μόνο με αλληλογραφία επικοινωνούν. Ε, υπάρχει λοιπόν βέβαια που κλέπτεται και η αλληλογραφία και όλες οι επικοινωνίες. Δεν υπάρχει ιατρική περίθαλψη. Μόνο τρεις-τέσσερις μέρες το χρόνο έχουν άδεια. Καταλήγουν να τρώνε χόρτα γιατί το φαΐ εκεί είναι πάρα πολύ κακό Οπότε πρέπει να φροντίσουμε πραγματικά ο ευρωπαϊκός πολιτισμός να μην ε, χρεωθεί το αίμα αυτών των ανθρώπων. Ευχαριστώ για ένα λεπτό κύριος Γκρίφιν. Η προοπτική της φυλάκησης ε, για εγκλήματα της σκέψης ουσιαστικά είναι αποτροπιαστική. Και είχα τέτοια εμπειρία γιατί τρεις φορές προσπάθησε η Βρετανική κυβέρνηση να φυλακίσει μόνο και μόνο επειδή είπε την αλήθεια. Αυτό όμω δεν είναι αδίκημα, παρόλο που επικαλέστηκε για διάφορα νομοθετήματα. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στην Κίνα. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να σταματήσουμε την εισαγωγή τέτοιων προϊόντων από στρατόπεδα Λαογκάι. Είναι καταναγκαστική αυτή η εργασία και η εισαγωγή τέτοιων προϊόντων συνιστά θέμη τον ανταγωνισμό. Μάλιστα, οι, κρατούμενοι αυτοί δεν μπορούν καν να συνδικαλιστούν, δεν υφίσταται καμία προστασία, καταπατούνται και περιβαλλοντικοί κανόνες. Η εισαγωγή τέτοιων προϊόντων συνιστά αθέμητο ανταγωνισμό. Επίσης, κατα... καταρακώνουν τον βιομηχανικό μας ιστό και τη μεταποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα πρέπει τέτοια προϊόντα κομμουνιστικής τυραννίας να έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. ένα λεπτό, συνάδελφος. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα πρέπει να διακρίνουμε τους κρατούμενους που έχουν διαπράξει κάποια δίκημα και τους πολιτικούς κρατούμενους. Τώρα, το εάν είναι σωστό το και δίκαιο το δικαστικό σύστημα καθώς επίσης και το εάν είναι σωστές συνθήκες στα λαογκάι. Το εάν επιτρέπεται όμως να τα αγοράσουν αυτά τα προϊόντα άλλοι άνθρωποι εξαρτώνται από το εάν η χώρα η οποία εισάγει θέλει να κλείσει τα δικά της εργοστάσια και να αφήσει τους ανθρώπους τους άνεργους. Αυτό ισχύει όχι μόνο σε αγαθά που παράγουν φυλακισμένοι, αλλά αγαθά παρόντα σε οποιαδήποτε χώρα με χαμηλού μισθού με του οποίου δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε. Βέβαια, ε, οι υπέρμαχοι του ελεύθερου εμπορίου λένε πω με το ελεύθερο εμπόριο γίνεται ο κόσμο πιο πλούσιο. Όχι όμω κάθε μεμονωμένη χώρα, ούτε οι Βρετανοί και οι Ευρωπαίοι άνεργοι. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μπρόνς. Τέλος έχει ο Επίτροπος ο κύριος Φίλιο τον λόγο πάλι. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη Ευρωβουλευτέ, η οικονομική ανάπτυξη της Κίνας είναι άνευ προηγουμένου στη σύγχρονη οικονομική ιστορία και παρόλο που και ταυτόχρονα διαδραματίζει όλο και σημαντικότερο ρόλο στην παγκόσμια οικονομία και σκηνή. Βέβαια, θα πρέπει ταυτόχρονα να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Η κινέζικη ηγεσία θα πρέπει οπωσδήποτε να τηρήσει αυτές τις προκλήσεις. Η Κίνα είναι φυσικό εταίρος Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο διάλογος με τη χώρα αυτή είναι ο καλύτερος τρόπος για να προσπαθήσουμε να διαθετήσουμε αυτά τα θέματα στα πλαίσια του διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά και στα πλαίσια του υψηλού επίπεδου οικονομικού και εμπορικού διαλόγου που έχουμε τη χώρα αυτή. Τούτου λεχθέντος θα πρέπει να εμείνουμε στις αξίες και τις αρχές μας και σε ό,τι αφορά την καταναγκαστική εργασία σε στρατόπεδα Λαογκάι. Όπως είπα και στην εισαγωγική μου ομιλία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται, είναι ανοιχτή να διερευνήσει αποτελεσματικούς τρόπους για να απαγορεύσει την εισαγωγή αγαθών που παράγονται με εργασία καταναγκαστική σε τέτοια στρατόπεδα. Και προσβλέπουμε σε στενό διάλογο για το θέμα αυτό με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο Επίτροπο Κάλντε Κούχτ αναφέρθηκε εκτενώς την περασμένη Τρίτη σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα. Σα διαβεβαιώ ότι το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα αποτελέσει μέρος της ημερήσιας διάταξης της ε, ε, διάσκεψη κορυφής της 6ης Οκτωβρίου με την Κίνα και θα προτείνουμε ακόμη και κατάργηση, κλείσιμο αυτών των στρατοπέδων Λαογκάη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως στερείται οριζόντιου μηχανισμού για την απαγόρευση τέτοιων αγαθών που παράγονται με την ε, εργασία των κρατουμένων. Πάντως, ε, πρόκειται να εξετάσουμε και την αποτελεσματικότητα του Αμερικανικού δικαίου για την απαγόρευση τέτοιων αγαθών, μια και είναι πολύ δύσκολη ανείχνευση της προέλευσής τους. Τέσσερις επίτροποι και οι αντίστοιχες γενικές διευθύνσεις ασχολούνται με το θέμα αυτό. Και σας διαβεβαιώ ότι και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ήρθε η ώρα να ενισχύσει την ε, συνεργασία μεταξύ των διαφόρων γενικών διευθύνσεων προκειμένου να βαθύνει στην ανάλυση του θέματος αυτού. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Εδώ πέρα τελειώνει η συζήτηση. Τα πρακτικά της χρησινής συζήτησης και τα κείμενα που ευθύθηκαν στη διάστηση των συναδέλφων υπάρχουν αντιρρήσει πρακτικά. Όχι, άρα τα πρακτικά εγκρίνονται. Κυρίε και κύριοι, σα ανακοινώνω πω η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων στι 20 Σεπτεμβρίου 2010